Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε ένα πόλεμο κατά της ομοφοβίας, κατά της αρνητικής αντιμετώπισης των ε, διεμφυλικών και μεσοφιλικών ατόμων. Σας διακόπτω, λέει η Πρόεδρος, έχουμε καθυστερήσει ήδη πολύ. Θα πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι ομιλητές. Η κυρία Ιντβέλτορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν από όλου του συναδέλφου, διότι Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Μερικά σχόλια για το τι κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όπως και οι συνάδελφοί μου, καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που έχουμε το πρώτο ψήφισμα στη ημερησία διάταξη για τα μεσοφιλικά άτομα. Μεγάλο, πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα ψήφισμα ε, για ε, τις ε, δράσεις ε, για τους ΛΟΑΔΜ που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή της θητείας. Και αυτά τα ψηφίσματα θα πρέπει να είναι μια κληρονομιά ε, προς ε, την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επόμενο Κοινοβούλιο όπου να ζητούμε πιο ισχυρή δράση από όσοι έχουμε αναλάβει την τελευταία πενταετία. Διότι πιστεύω ότι απομένουν πολλά να γίνουν. Βεβαίως έχουν επιτευχθεί πολλά στο ε, ε, Συμβούλιο, ας πούμε, σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις, τα κράτη-μέλη δεν ε, συμφώνησαν καν για μια κοινή δήλωση για τα δικαιώματα ΛΟΑΔΜΑ. Μα καλά στο μεσαίο να είμαστε ακόμα. Γιατί τα μπλοκάρουν τα κράτη και η οδηγία αυτή για τις διακρίσεις είναι σε εμπλοκή για μια δεκαετία και πλέον. Αλλά και εδώ στο Κοινοβούλιο, ο ίδιος ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ταγιάννη, είναι από τους βασικούς ομιλητές στο Παγκόσμιο Συνέδριο ε, Οικογενειών που είναι ε, από τα πιο ομοφοβικά πράγματα και εκδηλώσεις στον κόσμο και κατά της επιλογής σε μια οργάνωση που λέγεται Citizen Go που είναι ε, πρωταθλήτρια της λεγόμενης διακήρυξης του Νάσβιλ, που είναι η πλέον ομοφοβική παγκοσμίω. Και ορισμένοι εδώ μέσα την έχουν προσυπογράψει. Εγώ δεν θεωρώ ότι με εκπροσωπεί ο κύριο Σταγιάννη που εμφανίζεται σε μια τέτοια εκδήλωση και να έρχεται εδώ να ε, υποστηρίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ. Αυτό είναι ε, η υποκρισία πραγματικά σε όλο τη το μεγαλείο. Η κυρία Ρέντκε για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει ε, ισχυρά τις ε, χειρουργικές παρεμβάσεις ε, για υποτιθέμενη εξομάλυση του φύλου. Αυτό αλλάζει την ιστορία. Είναι ε, μια απλή δήλωση και συχνά απλέ δηλώσει είναι αυτές που αλλάζουν την ιστορία. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε ιστορία όταν θα ψηφίσουμε το πρώτο ψήφισμα για τα μεσοφιλικά άτομα εδώ στο Κοινοβούλιο. Και βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να ε, διορθώσουμε ε, όλα τα δεινά ε, που έχουν προκληθεί στις ζωές των ανθρώπων, αναγκαστική στήρωση, θεραπείες και χειρουργία παρά τη θέλησή τους, στιγματισμός και διακρίσεις. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε αύριο είναι να διατρενώσουμε ότι θα αγωνιστούμε για ένα μέλλον όπου τα δικαιώματα των μεσοφιλικών ατόμων θα διατηρούνται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Έπρεπε να το είχαμε στείλει νωρίτερα αυτό το μήνυμα, αλλά έρχεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Γιατί τα δικαιώματα όλων των ΛΟΑΔΜ αυτή τη στιγμή ε, διώκονται και πλήττονται. Μετά από δεκαετίε προόδου, τώρα κινδυνεύουμε να οπισθοδρομήσουμε. Για να το αποτρέψει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εγκρίνει μια στρατηγική ακριβώ για την πρόληψη, με ένα νέο κατάλογο δράσεων για του ΛΟΑΔΜ και τα δικαιώματά του. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ε, υψώσει το ανάστημά της ε, απέναντι σε εκείνους που δεν αφήνουν κάποιους άλλους να ζήσουν όπως θέλουν. Τι θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απεμπλακεί η οριζόντια οδηγία για την ισότητα ε, που έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο και στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας να δώσει συνέχεια για ελεύθερη κυκλοφορία των ΛΟΑΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των διακρίσεων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οφείλουμε αυτό στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνω το κατάλογο των ομιλητών και παρακαλώ τον Υπουργό, τον κύριο Τσάμπα, να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρία Επίτροπε. Να ευχαριστήσω καταρχά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δυνατότητα που μα δίνει να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα σήμερα εδώ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίω στα δικαιώματα των μεσοφιλικών ατόμων που θα πρέπει να προστατεύονται σε όλα τα κράτη-μέλη και αποτελούν βέβαια το αντικείμενο της ερώτησής σας προς το Συμβούλιο. Θα ξεκινήσω λέγοντας ξεκάθαρα ότι η βία και η διακριτική μεταχείριση δεν έχουν θέση σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θέσει την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης ως πρωταρχική προτεραιότητα. Οι αρχέ και οι αξίε Ευρωπαϊκή Ένωση, των συνθηκών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση. Στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών και την αξιοπρέπεια όλων των πολιτών. Μόνο έτσι θα έχουμε δίκαιε κοινωνίε. Αυτό ισχύει για όλου του Ευρωπαίου και βέβαια για ένα πολύ καλό λόγο. Οι κοινωνίες μας γίνονται κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Πολύ περισσότερο από ποτέ. Από κοινού λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ισότιμη μεταχείριση για τις γυναίκες και για όλες τις μειονότητες, σεξουαλικές μειονότητες, θρησκευτικέ μειονότητες, άτομα με αναπηρίες και ούτω καθεξής. Και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για το ζήτημα αυτό. Όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν ότι θα πρέπει αυτή την άγουσα να ακολουθήσουμε, μια μεγαλύτερη δηλαδή ανοχή για τα άτομα αυτά και μεγαλύτερη χειραφέτηση για αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Είμαι σαφώς υπέρ της προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση διακριτικής μεταρρύθμισης βάσει του άρθρου 19 της Συνθήκης και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν ορισμένοι λόγοι διακρίσεων που αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα σε ορισμένα κράτη-μέλη από ότι άλλοι λόγοι. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να σημειώσουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη βία και την διακριτική μεταχείριση για τα μεσοφιλικά άτομα. Όντω, αναφερθήκατε σε πραγματική οδύνη για τα άτομα αυτά. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την προφορική σα ερώτηση. Με ιδιαίτερη περηφάνεια πρέπει να πω, τον Ιούνιο του 2016 το Συμβούλιο ανταποκρίθηκε θετικά στην, στον κατάλογο δράσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθηθεί η ισότητα των ατόμων ΛΟΑΔΜ. Για πρώτη φορά το Συμβούλιο τότε ενέκρινε μία δήλωση όπου ρητά γίνεται αναφορά στην βελτίωση της ισότητας των λεσβιών, ομοφιλοφίλων, διεμφυλικών και μεσοφιλικών ατόμων. Η στιγμή αυτή λοιπόν τα πραγματικά ιστορική. Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει περισσότερο τα μέτρα αυτά τα οποία προβλέπονται στο κατάλογο δράσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ενημερώνει το Συμβούλιο τακτικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα έχει επιτύχει. Και μάλιστα καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη στα πλαίσια τη εθνική του νομοθεσίε και τη εθνική αρμοδιότητα να προωθήσουν περισσότερο στρατηγικές καταπολέμησης των διακρίσεων, αξιότιμα μέλη. Η πρόθεση τη ισότιμη μεταχείριση πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο όλων μα. Όσον αφορά τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κατάλογο δράσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, θα πρέπει να χαιρετιστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω έχει ξεκινήσει και μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης Επίση, ε, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει συμβάλει και αυτό πάρα πολύ, χαρτογραφώντα την κατάσταση των μεσοφιλικών ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την καταχώρηση γεννήσεων ή όσον αφορά τι περιπτώσει αναγκαστική χειρουργική επέμβαση, στην οποία αναφερθήκατε, ή όσον αφορά το ζήτημα τη ενεπιγνώση συνένεση. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με βασική ιατρική δοντολογία, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι εθνική αρμοδιότητα, για την οποία λογοδοτούν τα κράτη-μέλη. Το ζήτημα της καταχώρησης των γεννήσεων είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, που όμως και αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Προφανώς υπάρχει. Όπω ξέρετε, η κατηγορία των μεσοφιλικών ατόμων δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ε, περιπτώσεων εκείνων που θα πρέπει να απαγορεύονται συγκεκριμένε διακρίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε λοιπόν και αυτό το αίτιο και αυτή τη βάση, αν θέλετε, διακριτική μεταχείριση. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε τελικά να οδηγηθούμε σε κοινωνίε οι οποίε θα λειτουργούν χωρί αποκλεισμού. Καθώ προσπαθούμε να προωθήσουμε και να περασπίσουμε τι αξίε μα, Εποφελούμεθα όλοι από τις επικοδομητικές ανταλλαγές απόψεως απόψεων σαν αυτή που έχουμε εδώ πέρα σήμερα και η οποία θα επιβεβαιωθεί ακόμα περισσότερο από την αυριανή ψηφοφορία. Όπως σας είπα στην αρχή της παρέμβασής μου, η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα την καταπολέμηση διακριτικής μεταχείρισης και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και το λέω αυτό με ιδιαίτερη περηφάνεια. Σα ευχαριστούμε, Επίτροπο Γιούροβα, έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την ε, διενέργεια τη αυτή της συζήτησης ε, που κάνουμε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προσήλωση εργάζεται για την ε, προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΤΜ και χαιρετίζει το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο ε, πρόκειται να ψηφίσει ε, αυτή την έκθεση και διατηρεί ε, ψηλά στην λίστα των προτεραιοτήτων το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό ακριβώς δημοσιεύσαμε και εμείς τον κατάλογο δράσεων για την πρόθεση της ισότητας των ΛΟΑΔΜ το 2015. Τους επόμενους μήνες ε, θα παρουσιάσουμε και μια τρίτη έκθεση ως προς την ε, υλοποίηση ε, των ενεργειών που βρίσκονται στον κατάλογο. Θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα στο τέλος της παρέμβασής μου. Να σταθώ επιγραμματικά στα προβλήματα των μεσοφιλικών ατόμων που όπως ξέρουμε όλοι και υπόθηκε και πολλές φορές σήμερα, αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα γιατί δεν ε, εντάσσονται στις ε, κύριες ε, ταυτότητες φύλου του άντρα και της γυναίκας. Υπάρχουν λοιπόν περιτές, μη απαραίτητε χειρουργικές επεμβάσεις στα μεσοφολικά άτομα που είναι απαράδεκτες ακριβώς και επειδή είναι πολύ νέα αυτά τα άτομα όταν υφίστανται τις επεμβάσεις. Ο ορισμός των πολιτικών υγεία και τη διοργάνωση και παροχής υγειονομικών υπηρεσιών εμπίπτει ε, την αρμοδιότητα κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται την επικουρικότητα λοιπόν σε ό,τι αφορά την ε, νομική ευθύνη ε, για τις επεμβάσεις αυτές, σε ό,τι αφορά ανήλικους. Πρόκειται λοιπόν για αρμοδιότητε ε, των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τα διαφιλικά άτομα, τα κρατημέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι ε, τηρούνται οι απαραίτητε ε, και σχετικέ ρήτρε βάσει και των διεθνών προτίμων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε και επεφάνθη ότι ε, οι επεμβάσεις αυτές ε, ε, αντίκυνται στο άρθρο 8 της Σύμβασης. Επιστρέφω στο κατάργο των ενεργειών που έχουν ως στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων ε, των ΛΟΑΔΜ. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, υλοποιήσει μια σειρά ενεργειών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ό,τι φορά τις ε, συνθήκες ζωής αυτών των ατόμων. Δημοσίευσε πρόσφατα και μια μελέτη για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ και τα δικαιώματά τους στην Ευρώπη. Στηρίζουμε και ΜΚΟ και οργανώσει κοινωνία των πολιτών που προωθούν την ισότητα των ΛΟΑΔΜ και των μεσοφιλικών. Έχουμε δημοσιεύσει ορισμένα βίντεο ε, αύξηση τη ευαισθητοποίηση και έχουμε διοργανώσει και έναν ε, κοινωνικό διάλογο σε μια σειρά των μελών. Υπάρχει και το πολιτικό έργο για την υγεία των ΛΟΑΔΜ και πάλι με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που άπτονται της υγείας ε, των ΛΟΑΔΜ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον παρακολουθεί και ενισχύει ε, τα ισχύοντα δικαιώματα ε, με βάση τη σχετική οδηγία. Και χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση ε, του δικαστηρίου και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την συμμόρφωση των κρατομελών σε ό,τι αφορά το κεκτημένο για το ζήτημα αυτό θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τον κατάλογο ενεργειών για την προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και το 2019. Φέτος θα έχουμε και ένα νέο ευρωβαρόμητρο που θα περιλαμβάνει και ερωτήσεις για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ και θα γίνει και η δεύτερη ε, σχετική μελέτη που θα μας δώσει στατιστικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να στοχεύσουμε καλύτερα τις μελλοντικέ μας δράσεις. Είναι μια χρονιά αξιολόγησης και προπαρασκευαστικού έργου για την μελλοντική μελλοντικό αναθεωρημένο κατάλογο ενεργειών για τα άτομα ΛΟΑΔΜ που θα υιοθετηθεί από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο. Ε, θέλουμε και παλεύουμε να έχουμε προωθήσει αυτό το θεματολόγιο ε, όταν θα το παραδώσουμε στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως ε, σίγουρα θα μεταφέρω αυτό το μήνυμα και στον διάδοχό μου να λάβει υπόψη την προσέγγιση ΛΟΑΔΜ στην διαμόρφωση πολιτικής στο μέλλον καθώς και το σημερινό ψήφισμα. Να Κάνω και μία σημείωση για τη σημερινή συζήτηση. Εμείς θέλουμε την υιοθέτηση της ε, οριζόντιας ε, οδηγίας ε, ίσης μεταχείρισης. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι έχει μπλοκαριστεί εδώ και χρόνια αυτή η πράξη στο Συμβούλιο. Γνωρίζετε ότι η νομοθετική αυτή πράξη απαιτεί ομοφωνία. Γι' αυτό και πρέπει όλα τα κρατημέλη να συμφωνήσουν και είπα ότι μετά από τόσα χρόνια η συνθήκη ε, προσφέρει και την ε, ε, επιλογή της ενισχυμένης συνεργασίας και προς έκπληξή μου είδα ότι και στις συνδύσεις του Συμβουλίου και στις διμερείς συζητήσει, πολλά κράτη-μέλη είπαν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο και δεν θέλουν να ακολουθήσουν με την ενισχυμένη συνεργασία γιατί είναι ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ήθελα απλώς να το ε, μεταφέρω. Και θα συνεχίσω να ασκώ πιέσεις. σε ό,τι αφορά αυτή την οδηγία. Κάτι τελευταίο. Μιλήσατε και για ε, τη ρητορική μίσους και στο διαδίκτυο αλλά και εκτός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται με προσήλωση από κοινού και με το τομέα της πληροφορικής για να πετύχουμε δραστική μείωση της ρητορική του μίσους ε, στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με αρκετή επιτυχία. Ο τομέας της προφορικής ε, πράττει τα δέοντα με βάση και τον κώδικα δεντολογίας και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια σίγουρα μέχρι το τέλος της θητεία μου. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συνεχίζεται η συζήτηση. Το λόγο έχει ο κύριο Φαρία. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε, Επίτροπε. Μετά το κίνημα Me Too, χιλιάδες ΛΟΑΔΜΑ ε, έχουν βγάλει στο Twitter διάφορες ιστορίες για εκφοβισμό κτλ. Στον 21ο αιώνα δεν μπορεί να εμφίσταται διακρίσεις οι πολίτες και οι Ευρωπαίοι πολίτες λόγω ε, ε, της ταυτότητάς τους και ε, οι ΛΟΑΔΜΑ ακόμα δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δεν χαίρουν των ίδιο δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αναλάβουμε δράση και μέτρα για την προστασία τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ε, παιδεία, υγεία, ε, κοινωνική ασφάλιση. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς, μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναγνωρίζεται η ταυτότητα και των μεσοφιλικών ατόμων και να έχουμε στρατηγικές για την πρόληψη βίας ε, ομοφοβικής και τρανσφοβικής και μάλιστα και τα παιδιά τους να προστατεύονται. Ευχαριστώ η κυρία Γουόρντ. Όταν συζητούμε για ε, τους ανθρώπους ΛΟΑΔΜ, ξεχνάμε τα μεσοφιλικά άτομα εδώ και αιώνες ε, τους ε, είχαμε στερήσει την ανθρώπινη υπόσταση λόγω του σώματός του. Το θεωρούσαν πρόβλημα υγείας. Μα δεν υπάρχει θέμα υγεία στα μεσοφελικά άτομα. Ε, συνέχεια ακολούθησαν ε, αναγκαστικοί ακροτηριασμοί. Είναι φρικαλαιότητες αυτά και τελείως απαράδεκτα το 2019. Ε, συνεχίζονται αυτές οι παραβιάσεις της αυτονομίας του σώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίνουμε ε, να κάνουμε αυτή την αλλαγή σε παιδικά σώματα και μάλιστα μόνιμη και μη αντιστρεπτή. Ε, πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη γελία ε, αντίφαση μεταξύ ανδρών και γυναικών ή άντρα θα είσαι η γυναίκα. Τα μεσοφελικά άτομα έχουν αποδείξει ότι δεν μπορείς να ταξινομήσεις σε κατηγορίες με βάση ε, τα χαρακτηριστικά του φύλου. Ε, ε, αυτά είναι οι αγγελώσεις. Θέλω να πω στους ανθρώπους αυτούς τους μεσοφελικούς και ιδιαίτερα στα παιδιά, δεν είστε μόνοι σας. Η κυρία Στέβενς, για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ακόμα και Τώρα τα δικαιώματα των ε, ΛΟΑΔΜ δεν είναι εγγυημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Δεν έχουμε ενιαία συνολική προστασία κατά της διάκρισης με βάση την ταυτότητα του φύλου, το γενετήσιο προ... Ε, ε, συνανατολισμό ή τα χαρακτηριστικά του φύλου. Πολλά κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν τους γάμους μεταξύ δύο ανδρών ή δύο γυναικών, που στο Βέλγιο υπάρχει. Ακόμα 8 κράτη-μέλη ε, δέχονται τους ακροτηριασμούς και τη στήρωση, ενώ 18 κράτη-μέλη έχουν ψυχολογική βία. Ε, σε 21 κράτη στα μεσοφιλικά παιδιά κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις ε, δίθεν εξομάλυσης. Τι γίνεται με τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παραβιάζεται. Υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να θέσει προτεραιότητες στα δικαιώματα των ε, ε, ΛΟΑΔΜΟ για το 2019 2020 θα πρέπει να ενισχυθεί και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων έτσι ώστε τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΟ όπως είναι δικαίωμα στην υγεία και την παιδεία να ε, διαπερνούν όλε τις πολιτικές. Επίσης έχει σημασία η Ευρώπη να συνεχίσει τις εξαρτίε συνειδητοποίηση για του ΛΟΑΔΜΟ και τι οικογένειε του. Θα πρέπει επίσης η Ευρώπη να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των ζευγαριών ε, και ΛΟΑΔΜ. Ε, το έχουμε δει και πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τέλος, είναι απαράδεκτο η ΛΟΑΔΜ σε πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης να θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ένστ για 1,5 λεπτό. Σήμερα συζητούμε για πρώτη φορά ένα ψήφισμα για τα δικαιώματα των μεσοφιλικών ανθρώπων. Και πραγματικά έχει έρθει η ώρα. Γιατί έχει γίνει ταμπού αυτό το θέμα. Και διευκολύνει ε, το να βάζουμε κάποιους ανθρώπους να τους κλειδώνουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ε, της έλλειψης δικαιωμάτων. Και κάποιοι άλλοι αποφασίζουν τι είναι σωστό για αυτούς ότι θα πρέπει το λανθασμένο ή απόκληση να διορθώνεται εντό εισαγωγικών και με χειρουργική επέμβαση. Ό,τι και να λέμε σήμερα, ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον για το εξής. Θα πρέπει με κάθε δύναμη να φροντίζουμε τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις να απαγορεύονται στα νεογνά, στα βρέφη, παντού γιατί ε, δεν χρειάζονται για λόγους ιατρικούς. Δεν είναι άρρωστοι οι άνθρωποι μεσοφιλικοί που να χρειάζονται θεραπεία. Είναι φυσιολογικοί άνθρωποι που ε, θέλουν να αποφασίζουν για τον εαυτό τους και να τους σέβονται οι άλλοι. Κανένας δεν θα πρέπει να φοβάται ε, ότι θα το πιθαναγκάζουν, ότι θα το φημώσουν, ότι θα το κάνουν για να αμφιβάλλει για τον ίδιο του τον εαυτό θα πρέπει πραγματικά να διώκονται ποινικά αυτά τα πράγματα. Ε, ενημέρωση της κοινή γνώμης, θετική ενημέρωση και εξομάλυνση της συζήτησης. Τώρα το τι θα γράφουν οι ταυτότητες ή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι επιτέλους ε, η ανθρώπινη ζωή δεν είναι μονόδρομος. Ευχαριστώ κύριος Λόπες Ακυλάρ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, Επίτροπε Γιώροβα, ένα ηθικό ζήτημα, ε, μάλλον ε, μια, ένα προφορικό ερώτημα, είναι κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ψηφίσουμε την Πέμπτη. Εγώ έχω συμμετάσχει σε όλε τι ε, συζητήσει σχετικά με την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πιο ευάλωτων ομάδων. Περί αυτών πρόκειται. Έχουν υποστεί τεράστιες διακρίσεις, ακόμα και ποινικοποίηση και ποιος αποφασίζει για αυτός. η ΛΟΑΔΜ, η ε, ε, διεμφυλική και η μεσοφυλική ε, υποφέρουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και να τις ακολουθήσουμε. Τα μεσοφιλικά άτομα, η, η γενετήσια προτιμήση δεν θα πρέπει να θεωρείται αρρώστια και να προσπαθούν να τους γιατρέψουν με τρόπο χειρουργικό ή φαρμακολογικό. Θυμάστε το 2014 ψηφίσαμε την έκθεση Λούνατσεκ για μια θεώρηση συνολική και χωρίς αποκλεισμού των δικαιωμάτων. Ε, και ο πρόεδρο, η πρόεδρος διακόπτη τον ομιλητή, ζητώ συγγνώμη, θα πρέπει να τηρείτε το χρόνο σας. Κάτι στη θα έχουμε για αυτή τη συζήτηση, αλλά έχουμε καθυστέρηση 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και θα πρέπει ε, να τη μειώσουμε αυτή. Η κυρία Φορένζα, για ένα λεπτό ακριβώς παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι διεξάγεται αυτή η συζήτηση από κοινού για τα μεσοφιλικά άτομα και εν γέννη για τα άτομα ΛΟΑΔΜΑ και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε και ένα ψήφισμα όσον αφορά τα μεσοφιλικά άτομα. Όπως είπε ο συνάδελφος Βιώτη πριν από λίγο, νομίζω ότι τα όσα συζητάμε σήμερα και αν έχουμε σημειώσει πρόοδο, το οφείλουμε τελικά σε όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στη διακομματική ομάδα για τα άτομα ΛΟΑΔΜΑ, στην οποία συμμετέχω και εγώ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε και ένα κίνημα φεμινιστικό, το οποίο όλο και περισσότερο παρουσιάζεται ως τρανσφεμινιστικό κίνημα, καθότι δεν επικεντρώνεται μόνο στη χειραφέτηση των γυναικών, αλλά στην απελευθέρωση και χειραφέτηση όλων των ατόμων ΛΟΑΔΜΑ. Θα πρέπει να καταδικάσουμε οποιαδήποτε μορφή χειρουργικής επέμβασης που γίνεται στα παιδιά, τα μεσοφιλικά, προκειμένου να τους δοθεί το ένα ή το άλλο φύλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν για τη σημερινή συζήτηση που διεξάγουμε εδώ. Ευχαριστούμε κύριο Σάτσνατς. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανησυχεί για τα άτομα αυτά τα οποία έχουν σεξουαλικές δυσλειτουργίες, τα αποκαλούμενα ΛΟΑΤ, ΜΛΟΑΤ και δεν ξέρω και εγώ τι. Νομίζω ότι παρασχολούμεθα με τους ανθρώπους αυτούς και ξεχνάμε άλλα σημαντικά ζητήματα των κοινωνιών μας και μάλιστα έχουν και πολλά προνόμια άνθρωποι αυτοί γιατί πρόσφατα στο Μένο Βασίλειο είχαμε μια κατάσταση όπου, μια, όπου η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα στο σπίτι της γιατί μέσω διαδικτύου αποκάλεσε έναν άνδρα άνδρα, ενώ ο άνδρας αυτός είχε κάνει επέμβαση και είχε αλλάξει φίλο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και εγώ στο διαδίκτυο, οποιοδήποτε άλλο πολίτη να μπορούμε ελεύθερα να εκφράζουμε την άποψή μας. Νομίζω ότι αυτό που κάνετε εσείς και οι αριστεροί εδώ πέρα είναι ότι εκφοβίζετε τους υπόλοιπους πολίτες και προσπαθείτε ουσιαστικά να μειώσετε οποιαδήποτε επικριτική άποψη θέλουμε να εκφράσουμε. Κυρία Γιούροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, εξαιρετικά μέλη. Μακρηγόρησα πριν, επομένω ε, θα είμαι πολύ συντομή τώρα. Να σας ευχαριστήσω για την ε, συζήτηση. Το Κοινοβούλιο και πάλι έδειξε μεγάλη προσήλωση ε, σε αυτό το θέμα. Το ίδιο κάνω και εγώ. Θέλω να εκφράσω τη βούλησή μου να εργαστώ για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Κάτι μπορώ να σας πω πιο συγκεκριμένα είναι ότι από κοινού με την διακομματική ομάδα ΛΟΑΔΜ θα πρέπει κάπως να εξολογήσουμε τον κατάλογο των ενεργειών, ε, κατά πόσο υπάρχουν ε, θετικά αποτελέσματα, αν πρέπει να αλλάξει κάτι στο μέλλον, στο επόμενο ε, σχέδιο δράσης ΛΟΑΔΜ. Θα έχουμε και νέα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συναντηθούμε και να εργαστούμε από κοινού. Αυτή είναι μια πρόσκληση λοιπόν που απευθύνω προς εσάς θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συνεργαστούμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο. Τέλος, ε, ο κύριος Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την ανταλλαγή απόψε. Νομίζω ότι από αυτήν προκύπτει ε, πόσα μένουν ακόμα να γίνουν. Παράλληλα, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τα βήματα που έχουμε σημειώσει σε αυτόν τον τομέα το Συμβούλιο ανταποκρίθηκε θετικά στη, στον κατάλογο ενεργειών ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την κοινότητα ΛΟΑΔΜ και προσβλέπω ε, στην περαιτέρω υλοποίησή του σε ό,τι φορά την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, βλέπουμε ότι η Ευρώπη είναι στην, ακολουθεί τη μεριά ε, της προόδου, της ανοχής και του φωτός. Είναι αρμοδιότητα των πολιτικών μας να μετατρέψουν ε, τις ε, προθέσεις σε πράξεις. Ευχαριστούμε. Έξι προτάσεις ψηφίσματος για να κλείσουμε αυτόν τον ε, διάλογο, μία από την Επιτροπή Λίμπε και μία από τις πέντε πολιτικές ομάδες. Η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καθώς περνούμε στο επόμενο σημείο τη μέση διάταξη που είναι προφορικό ερώτημα για τη χρήση τη Κάναβη για ιατρικού σκοπού, η οποία απευθύνεται προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνω ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία Catch the Eye, γιατί υπάρχει σημαντική υπέρβαση χρόνου. Ε, καταλαβαίνω ότι θα απογοητεύσω έτσι κάποιου συναδέλφου, αλλά με έχουν ενημερώσει ότι θα υπερβούμε ε, το χρονικό περιθώριο που είχαμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν, δεν ήμουν εγώ στο Προεδρείο προηγουμένω. Η κυρία Σουίτσα έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε πολύ με την υγεία, με την πρόσβαση στα φάρμακα, με τις υπηρεσίες υγείας κτλ. Και υπήρξε και προφορική ερώτηση ε, για τη χρήση της κάναβης για ιατρικούς σκοπούς. Τι ε, επιθυμούμε να βασιστούμε στη ε, χρήση επιστημονικών δεδομένων για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε την κάναβη για ιατρικούς σκοπούς. Η ιατρική κάναβη αποκλειστικά είναι το θέμα μας ε, και τίποτα άλλο. Υπάρχουν κείμενα που χωρούν ερμηνείες βέβαια ε, και δεν είναι ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε από τη μια τη χρήση της κάναβης για ιατρικούς σκοπούς και από την άλλη κάποιες καταχρήσεις που μπορεί να σημειωθούν ε, σε ό,τι αφορά τη χρήση της κάναβης γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να ε, ε, προβλέπουμε τη μέγιστη ε, συγκέντρωση THC στο κάθε προϊόν και κάθε κράτος μέλος να μπορεί να νομοθετεί για τα φάρμακα που έχουν κάναβη έτσι ώστε αυτά να μην χρησιμοποιούνται για αλότριους σκοπούς και να προκαλούν προβλήματα στους ασθενείς. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ε, εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ε, φρονεί για τη χρήση αυτών των ουσιών, σε ποια επιστημονικά στοιχεία βασίζεται και ποιες είναι οι έρευνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρηματοδοτήσει την έρευνα για τη χρήση κάναβης για ιατρικούς σκοπούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ε, δημιουργήσει κανόνες και πρότυπα για τη χρήση της κάναβης για μη ιατρικούς και μη φαρμακευτικούς σκοπούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές για ένα πάρα πολύ σαφή ορισμό της ιατρικής κάναβης καθώς επίσης και των τιμών και των ορίων ε, που θα πρέπει να περιέχουν τα φάρμακα. Ε, ε, θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση ανάμεσα σε φάρμακα που περιέχουν κάναβη και δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίες και εκείνα που κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται. Είναι πολλά τα μόρια καναβιοειδών, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και θα πρέπει να ε, κάνουμε διάκριση πραγματικά μεταξύ των ουσιών. Υπάρχουν πολλά φάρμακα τα οποία ε, πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένη δόση. Και ποιος θα επιφορτιστεί με την παραγωγή και ποιος θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο όλων αυτών των στοιχείων. Η πρόσβαση στα φάρμακα αυτά θα είναι ανοιχτή και για ανήλικες και ε, για ασθενείς που έχουν ειδικέ ανάγκες. Τι γίνεται με τις εγγύους, για παράδειγμα. Υπάρχει στην επιστημονική βιβλιογραφία αναφορά σε τέτοια χρήση κανάβεως. Υπάρχουν θεραπείες που απαιτούν αυτά τα φάρμακα όπως κάποιοι καρκίνοι, επιληψία, το άσθμα, άλλες χρόνιες παθήσεις. Υπάρχουν ε, ε, ασθένειες που προκαλούν σπασμούς ή υπάρχουν ασθενείς με χρόνιες ε, αγωνίες, κρίση πανικού ή κατάθλιψη. Θα πρέπει λοιπόν τα ερευνητικά κέντρα να προχωρούν σε ορισμούς σαφείς όλων αυτών των παθήσεων και των φαρμάκων και να χρησιμοποιούν τα φάρμακα αυτά μόνο οι ασθενείς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Ε, υπάρχουν ε, καθηγητές ε, και διάφοροι ακτιβιστές ε, που προσπαθούν να διαφημίσουν τη χρήση της καναβές. Όχι, θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρά, πλαισιωμένη και ρυθμισμένη η χρήση αυτή, αυστηρά η ιατρική χρήση, για να αποφευθούν ε, οι καταχρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Η Επίτροπος Γιώργο έχει το λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, την τελευταία δεκαετία είδαμε ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον του κοινού όσον αφορά τις θεραπείες που μπορούν να βασιστούν στην κάναβη και στα συστατικά της στοιχεία και αναφέρομαι όλο και περισσότερο, αναφέρεται η κοινή γνώμη και περισσότερο στην κάναβη γιατρική χρήση. Η θεραπευτική δράση της κάναβης έχει συζητηθεί για πάρα πολλές ασθένειες όπως η σκλήρηση καταπλάκας ή το άγχος ή το μετατραυματικό στρες. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διάκριση ανάμεσα στην μη φαρμακευτική ιατρική κάναβη καθώς επίσης και τα ιατρικά αυτά προϊόντα τα οποία μπορεί να βασιστούν στην κάναβη. Όσον αφορά τώρα το ρυθμιστικό πλαίσιο, η άποψη Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμοδιότητα μάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περιορισμένη. Μιλάμε πάλι εδώ πέρα για εθνική αρμοδιότητα. Κάθε εθνική φαρμακευτική αρχή τελικά θα πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να νομοποιήσει την κάναβη στην επιμέρους εδαφική επικράτεια. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι Προβλέπετε αυτή τη στιγμή σε ορισμένε χώρε να χρησιμοποιείται η κάναβη στα πλαίσια φαρμακευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμω θα πρέπει να έχει αποδειχθεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τη που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν. Αυτή τη στιγμή διατεθεί στην αγορά το φαρμακευτικό αυτό προϊόν, εξακολουθεί και παρακολουθείται μέσω δραστηριότητων φάρμακοεπαγρύπνησης, και αυτό ισχύει και για τα ιατρικά αυτά προϊόντα τα οποία βασίζονται στην κάναβη. Πώ μπορεί λοιπόν να συμβάλλει στη ζήτηση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία πρώτερη συζήτηση που έχει γίνει, καθώς επίσης και οι ιατρικές πυρογνωμοδοτήσει για τα ζητήματα αυτά μπορούν να συμβάλλουν πολύ. Μπορούμε να πετύχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να απαντήσω τώρα στο καθένα από τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Καταρχά, να τονίσω ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των καναβινοειδών και των σχετικών θεραπείων. Ευκαιρίε να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε περισσότερο την έρευνα αυτή θα προβλέπονται όλο και περισσότερο στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020. Καθώς επίσης και στο τελευταίο πρόγραμμα έρευνας είχαμε ανάλογες έρευνες. Πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στο παρελθόν όσον αφορά την έρευνα για την κάναβη και τα καναβινοειδή και τα άλλα συστατικά στοιχεία. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουμε την προσέγγιση αυτή και στο μέλλον. Στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο, το Horizon Ευρώπη, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την έρευνα συμπεριλαμβανομένων κάποιων καινοτόμων ε, τομέων που αφορούν και την θεραπεία. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, Πρέπει να σας πω ότι τα ζητήματα της οικονομικής περιθάλψης είναι περίπλοκα και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από τα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τα φαρμακευτικά προϊόντα προβλέπει την άδεια φαρμακευτικών προϊόντων που προβλέπονται από την κάναβη όταν τα προϊόντα αυτά έχουν αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση κανάβιος για ιατρικού σκοπού αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμβάλλει στην όλη συζήτηση. Τον Οκτώβριο του 2016 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας ξεκίνησε μία νέα έρευνα για την κάναβη που μας δίνει περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τη χρήση της ουσίας αυτής. Και το Δεκέμβριο του 2018 η υπηρεσία αυτή εξέδωσε μία μελέτη όσον αφορά την ιατρική χρήση της κάναβης και των καναβινοειδών. Και αυτό μπορεί να συμβάλλει σαφώς στην κατάρτιση εθνικών πολιτικών. Και κατά αυτόν τον τρόπο η υπηρεσία αυτή έχει συμβάλει στην όλη συζήτηση που διεξάγεται. Όσον αφορά τώρα την τρίτη ερώτησή σας, θα ήθελα να τονίσω ότι η μη φαρμακευτική ιατρική κάναβη βρίσκεται εκτός αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωση. Παράλληλα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι διεξάγεται παγκοσμίω μια συζήτηση, ιδίω στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Επιτροπής Τοξικονομίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά την αδειοδότηση, τη χρησιμοποίηση ψυχοδραστικών ουσιών. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής αυτής θα ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της φαρμακοιατρικής νομοθεσίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ιατρική χρήση της καναβέως έχει νόημα τα προϊόντα της καναβής μπορούν να βοηθούν τους ασθενείς, τους οποίους δεν πιάνουν τα άλλα φάρμακα. Στη συζήτηση αυτή, όμως θα πρέπει να προσέξουμε από δύο ακραίες καταστάσεις. Η πρώτη ακραία κατάσταση είναι όπως με το σκυλί του Παυλόφ. Ακούς κάναβη και αντιδράς. Αμάν, επικίνδυνο, τρομερό, παράνομα ναρκωτικά και θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι. Αλλά για τη φαρμακευτική ιατρική χρήση της κάναβης δεν ισχύει αυτό το αντανακλαστικό του Παυλόφ. Από την άλλη όμως θα πρέπει να προσέξουμε οι ασθενείς να μην ε, ε, θεωρούν αυτό που μου είπε ένας ασθενής, εγώ που είμαι γιατρός, ότι για να περάσει πλάτη μου πρέπει να καπνίσω ένα μπάφο, ένα και αλλιώς δεν μου περνάει. Ε, όχι. Δεν είναι για τους πόνους στην πλάτη. Ε, αυτά θα πρέπει να τα έχουμε σε ένα πλαίσιο ε, κανονιστικό, κανονισμένο, προσεκτικό και συμφωνώ απολύτως με την παράγραφο 14 ε, του ψηφίσματος, όπως να εγκρίνεται όπως και όλα τα άλλα φάρμακα δεν μπορούμε να βάζουμε τόσους περιορισμούς αλλού στη βιομηχανία και να πούμε για την κάναβη πάτε σκύλια λέστε. Ε, ελπίζω αύριο να το υποστηρίξετε με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μπαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εγώ είχα νομικό πόνο μια μέρα και στη Γαλλία πήγα να δω έναν νευρολόγο. Το μόνο που μου είπε είναι ε, καπνίστε ένα τσιγάρο. Το πρόβλημα είναι ότι αρχικά το κάπνισμα βλάπτει την υγεία και δεύτερον η κάναβη απογορεύεται στη χώρα μου. Μην νομίζετε ότι σε όλη την Ευρώπη μπορεί κανείς να ε, χρησιμοποιεί την ε, ε, ιατρική κάναβη. Δεν ισχύει αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να μας δώσει και να δώσει στα κράτη-μέλη σαφείς κατευθύνσεις. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το ψήφισμα που παρουσιάζεται εδώ είναι σαφές ότι πρώτα απ' όλα μέσω τη συνταχογράφηση ε, θα ελέγχεται αυτή η διαδικασία και είναι πολύ σημαντικό ε, ότι μόνο ο ιατρός είναι αυτός που μπορεί να συνταγογραφήσει την ιατρική κάναβη. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει και να την αγοράσει. Ε, την συνταγογραφή στο πλαίσιο συγκεκριμένων πόνων για τους ασθενείς. Όμως, Υπάρχει και μία σειρά τροπολογιών που έχουν κατατεθεί από τους συντηρητικούς ευρωβουλευτές που θεωρούν ότι μόνο η θεραπευτική μορφή ε, θα πρέπει ε, να θεωρείται χρήσιμη. Δεν ισχύει όμως, γιατί υπάρχει και μορφή ε, ήπιων συνταγογραφούμενων ουσιών που μπορεί να είναι πολύ πιο στοχευμένη και αποτελεσματική για συγκεκριμένους ασθενείς που δεν ανέχονται, αν θέλετε, δεν ανέχεται ο οργανισμό του τα, φάρμακα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα, να δώσουμε τη δυνατότητα στου γιατρού να, ε, να ακολουθούν και άλλε μορφέ θεραπεία που είναι πιο κατάλληλε για συγκεκριμένε ε, παθολογίε και προσωπικότητα. Δεν χρειάζεται να, να το κάνουμε ολόκληρο ζήτημα. Εδώ πρόκειται για την ε, θεραπευτική καναβή έτσι κι αλλιώς, ε, για τα μόρια CBD και δεν πρόκειται για την ε, ψυχολογική χρήση, το διευκρινίζω. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί λοιπόν εδώ, γιατί δεν χρειάζεται πάντα να κρύβονται τα φαρμακευτικά λόμπι από πίσω. Thank you for... Ευχαριστώ για ένα μισή λεπτό. Κρούπα. Στηρίζω όχι μόνο την έρευνα για νέα, ε, νέες αγωγές ε, φυσικής προέλευσης που έχουν λιγότερες ε, δυσμενείς παρενέργειες, αλλά και την πρόληψη που σχετίζεται περισσότερο με την περίθαλψη και θα εξαλείφει παράγοντας κινδύνου. Βλέπουμε στο ψήφισμα ότι τα επίσημα στοιχεία για την έρευνα και χρηματοδότηση της ιατρικής κάναβης είναι σχεδόν ανύπαρκτη οι συνέπειες χρήσης ε, των προϊόντων κάναβης αφορούν μόνο πολύ συγκεκριμένες ε, δράσεις και θετικές ε, επιπτώσεις μετά από θεραπεία. Πρέπει λοιπόν πρώτα να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα για τον αντίκτυπο των ουσιών CBD πριν εισαγάγουμε γενικευμένη χρήση της κάναβης. δεν φαίνεται πολύ ε, σόφρον να έχουμε ε, την ε, γενικευμένη αγωγή κάναβης. Πρώτα πρέπει να έχουμε τις κλινικές δοκιμές και μόνο μετά να περάσουμε σε αγωγές. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει μόνο αν τα ωφέλη υπερτερούν των παρενεργειών και βλέπουμε ότι σε πολλές ασθένειες ε, χρησιμοποιούνται αγωγές ε, ε, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα ερευνητικά στοιχεία. Ιδίω σε συγκεκριμένε περιπτώσει που χρειάζεται όλα ένα για μεγαλύτερη δόση. Ο κύριο Φλάνναγκαν. Υποστηρίζω τα περισσότερα από το ψήφισμα αυτό. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο για να υποστηρίζουμε την νομιμοποίηση της ιατρικής κάναβης παντού θα πρέπει να τερματιστεί η κατάσταση. Ε, όπως κάποιοι γνωστοί μου που έξι φορές ε, το χρόνο πηγαίνουν στις κάτω χώρες για να βρουν το φάρμακο για την κόρη τους θα πρέπει να μπορεί να εισάγεται αυτό το αποδεδειγμένο φάρμακο και να τους το δίνουν στο σπίτι τους, να τους το ε, παραδίνουν. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ακρογωνιαίος λίθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας γίνει ε, ε, πραγματικότητα αυτό. Η Βέρα Τούμι και ο άνδρας της Οπόλ έχουν αποδείξει ότι μπορεί να βοηθήσει η κάναβη. χώρα της ε, ε, η κόρη τους είναι 9 χρονών και δεν χρειάζεται να τρέχει συνέχεια στο νοσοκομείο. Ε, θα πρέπει το φάρμακο αυτό να δίνεται σε όποιον τον έχει ανάγκη και ελπίζω να βοηθήσει το ψήφισμα στην κατεύθυνση αυτή. Η Επίτροπος, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση και ε, σύντομα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες που θα αυξήσουν τα επιστημονικά δεδομένα ε, και την επικοδομητική παροχή συμφουλών. Ευχαριστώ. Ε, λίγη εδώ η συζήτηση. Έχουμε λάβει μια πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και προχωρούμε τώρα στην προφορική ερώτηση με θέμα την γονιδιωματική τροποποίηση ανθρωπίνων ε, κιτάρων της βλαστικής σειράς. Θα δώσω το λόγο στον συντάκτη, κύριο Μικολάσιτς, για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το ζήτημα το οποίο υποβάλλουμε αυτή τη στιγμή προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαιρετική σημασία όχι μόνο για την μελλοντική εξέλιξη τη κοινωνία μας, αλλά και για την εξέλιξη του ίδιου του ανθρώπου, του ανθρώπινου είδου. Το γονιδίωμα των ανθρωπίων γεννητικών κυτάρων δεν έχει να κάνει μόνο με μια πολύ περιορισμένη πλεονέρευνα, έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στην επεξεργασία του γονιδιώματος μπορεί πραγματικά να οδηγήσει στη θεραπεία πολλών ασθενειών. Τούτο λεχθέντον όμως θα πρέπει να γίνεται μία διάκριση ανάμεσα στην επεξεργασία του γονιδιώματος των γεννητικών κυτάρων και του γονιδιώματος των σωματικών κυτάρων. Η επεξεργασία γονιδιώματος γεννητικών κυτάρων μπορεί να έχει πολύ επιβλαβείς επιπτώσεις. Μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές τροποποιήσεις οι οποίες θα περάσουν από τη μία γενιά στην άλλη και οι οποίες θα είναι μη αναστρέψιμες. Πρόσφατα είδαμε ότι ο Κινέζος ερευνητής Χεν Τσανκούι ανέφερε στην πρώτη κλινική χρήση της επεξεργασίας του γονιδιώματος γεννητικών κυτάρων και ε, ισχυρίστηκε ότι η επεξεργασία αυτή κατέληξε στη γέννηση δύο βρεφών. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Νομίζω ότι ε, εδώ πραγματικά θα πρέπει να δούμε ποια πρότυπα μπορεί ποτέ να ισχύουν πρότυπα ασφαλείας για αυτά τα γενετικά τροποποιημένα εντό αγωγικών μωρά. Το ζήτημα λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς αλλά και το τι ακριβώς έγινε. Η επεξεργασία του γονιδίωματο των γενετικών κυτάρων που μπορεί να είναι και κληρονομήσιμη ξέρει ότι αποτελεί αντικείμενο απαγόρευση. Υπάρχει σαφώ αναγνωρισμένη απαγόρευση διεθνώ για εντροποποίηση των γενετικών κυτάρων των ανθρώπων. Αυτή ακριβώ η επεξεργασία θέτει πολλού κινδύνου και θέτει επίση και πολλά ζητήματα τα οποία είναι διοντολογική φύση. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε ελαφρία την καρδιά ή να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό ή ότι θα δεν μπορούμε να αφήσουμε το ζήτημα αυτό μόνο στα χέρια των επιστημόνων και της, επιστημή... της επιστήμης. Χρειάζεται να δεξαχθεί μια πολιτική ευρεία συζήτηση που να βασίζεται σε συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία και να εμπλέκει όλη την κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθηθεί όλο και περισσότερο από το συμβόλο, Συμβούλιο μια απαγόρευση της τροποποίησης των γεννητικών κυτάρων και θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα για την περαιτέρω συζήτηση του ζητήματος αυτού. Σας ευχαριστούμε. Ο Υπουργό Τσάμπα έχει το λόγο, εξ ονόματος Συμβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, εξωτήμα μέλη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα μέλη σας για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα και να ευχαριστήσω τα δύο αξιότιμα μέλη που παρατήμασαν το προφορικό ερώτημα. Είναι γνωστή η προσήλωσή μας ε, στο ζήτημα των δεντολογικών συνεπειών που προκύπτουν από την αυξημένη γνώση που έχουμε του ανθρώπινου γονιδιώματος. Ε, γνωρίζουμε τις ε, πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις που αναφέρεται στο ερώτημα και που προκάλεσε γενική ανησυχία και προβληματισμό για τις συνέπειες προκύπτουν από τη δυνατότητα τροποποίησης του ανθρώπινου γονιδιώματος. Οι πρώτες δύο κλινικές δοκιμές με τροποποίηση του γονιδιώματος έχουν χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία ατόμου που ε, πάσχει από σοβαρή ε, ασθένεια. Κατανοούμε ότι η αυξημένη, η αυξανόμενη γνώση του ανθρωπίνου γονιδιώματος και των γενετικών αιτίων ε, ασθένειας μπορούν να συμβάλλουν στην, ε, ε, στο να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο σε αυτές τις σοβαρές ασθένειες. Από την άλλη πλευρά, μας προβληματίζει όλους ο κίνδυνος που μπορεί να ενέχει η τροποποίηση του γονιδιώματος στο μέλλον. Και υπενθυμίζω ότι η συζήτηση για τι εντολογικές συνέπειε της γνώσης σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα τροποποίησης ε, ε, του ανθρωπινού γονιδιώματος είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και με μερικές δεκαετίες. Πολιτικοί και επιστήμονες ε, έχουν επίγνωση της κατάστασης. Αυτό έχει οδηγήσει σε νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες για την σαφή ρύθμιση σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο γονιδίωμα και την ε, ε, αποτροπή της τροποποίησης ανθρώπινων γεννητικών κυτάρων. Σας ε, παραπέμπω και στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, ιδίω ό,τι αφορά τι φαρμακευτικέ ουσίε και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που απαγορεύουν την τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυτάρων. Σε ευχαριστώ την προσοχή στην στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ως πρώτη αρχή θέτει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απαγορεύει ρητό τέτοιου είδου ε, ε, πρακτικές ε, στον τομέα της ιατρική και της βιολογίας. Εξ όσων γνωρίζω, η τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυτάρων στην οποία αναφέρονται τα εξωτήμα μέλη είναι παράνομη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κατανοώ ότι ή ερμηνεύω το ερώτημά σα ως ένα απευθυνόμενο προς το μέλλον. Και η συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άρθρο τη συγκεκριμένα αναφέρει, ότι τα κράτη-μέλη έχουν ε, την ευθύνη ε, σε ό,τι αφορά την ιατροφορμικευτική περίθαλψη και είναι κάτι το οποίο λοιπόν θα πρέπει να ρυθμίζεται σε επίπεδο κράτου μέλου. Είμαι πεπισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το αποκλειστικά το δικαίωμα πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την ενωσιακή νομοθεσία. Και είμαι σίγουρος ότι παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ το ζήτημα. Αν θεωρείς ότι είναι ε, απαραίτητο, ε, θα προετοιμάσει τι ε, κατάλληλες νομοθετικές πράξεις. Και η Ρουμανική Προεδρία, αλλά και οι επερχόμενε προεδρίε. Ε, με τα χαρά θα εξετάσουν ε, τυχόν τέτοιες ε, προτάσεις. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ η επίτροπο. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση των διαδολογικών και νομικών ζητημάτων στις πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την γονιδιωματική τροποποίηση ανθρωπίνων πλαστικών σύρων. Γίνεται συζήτηση με διεθνείς οργανισμούς ε, για τη βιοιατρική και μια ε, ομάδε εργασία του ΟΣΑ για την βιοτεχνολογία, την νοτεχνολογία και συναφείς τεχνολογίες. Ε, συνεχίζεται λοιπόν σε ένα διεθνές επίπεδο αυτή η συζήτηση. Ε, είμαστε προσιλωμένοι μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επιβλέπουμε αυτές τις δραστηριότητες στο πρόγραμμα πλαίσιο της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία και τις κλινικές δοκιμές, καθώς επίσης και νομοθεσία για τα ιατρικά προϊόντα, ε, προβλέπουν ειδικέ διατάξεις που απαγορεύουν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα στιβαρό ρυθμιστικό πλαίσιο για ε, ιατρικά προϊόντα που υποστηρίζεται από τις αρχές της Σύμβασης του Οβιέδο ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων στη βιοιατρική. Ο κανονισμός 3094 το 2007 προβλέπει αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας ε, υγιεινής και ένα σύστημα συγκεντρωτικό για την έγκριση και την άδεια κυκλοφορίας. Ωστόσο, η απόφαση για τέτοιου είδου τεχνικές, για την, ε, τη γονιμοποίηση, η γονιμοποίηση, την εξωσωματική in vitro, ε, παραμένει ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με εθνικές αρχές για να ενισχύσουμε την, τον έλεγχο στις νέες τεχνολογίε τεχνολογίες στον κλάδο των ιστών και των κιτάρων. Η δεοντολογία ε, συνδέεται με τις νέες τεχνολογίες και αρμόδιες επιτροπές εξετάζουν μεταξύ άλλων ε, τις δεντρολογικές επιπτώσεις της γονιδιωματικής τροποποίησης ανθρωπίνων ε, γεννητικών κοιτάρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί διεθνώς τις εξελίξεις, τις δημοσιεύσεις και βεβαίως δεν είμαστε αντίθετοι στις νέες τεχνολογίες για ιατρικούς σκοπούς διοργανώνουμε και αντίστοιχη εκδήλωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Σας θυμίζω ότι δεν υπάρχει κατσιά εδώ και όλοι οι μελητές έχουν ένα λεπτό. Κύριε Λίζε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η σύγχρονη γενετική τεχνολογία δίνει καταπληκτικές ευκαιρίες που πρέπει εμείς να τις αδράξουμε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και δεοντολογικά όρια που θα πρέπει να τα σεβόμαστε. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε ό,τι είναι τεχνολογικά δυνατό. Ε, ο ερευνητής παρουσίασε στο Χονγκ κάποια αποτελέσματα ανεύθυνα. Όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι ε, επεμβάσει στην ανθρώπινη βλαστική σειρά είναι απαράδεκτέ και πρέπει να απαγορεύονται. Και χαίρομαι που γνώρισε και μεγάλη καταχραυγή στην επιστημονική κοινότητα, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί, να τραβήξουμε κόκκινε γραμμέ, οι οποίε να τηρούνται κιόλα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω ρητά το Συμβούλιο για την ε, ερμηνεία του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που θεωρώ το σωστή, αλλά θα πρέπει αυτό να μπει και στα μυαλά των ανθρώπων και στην νοοτροπία ότι αυτή η κατάχρηση απαγορεύεται. Θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού στην κατεύθυνση αυτή για να μην έχουμε επανάληψη τέτοιο φαινομένου. Ευχαριστώ. Κύριος Μπαλάς. Ε, μάλιστα. Ας είμαστε αυστηροί ε, το πρώτο στοιχείο είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι γίνεται ακριβώς με τις έρευνες που έκανε αυτός ο, ο Κινέζος επιστήμονας. Τίποτα δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά σε σχέση με τις ανακοινώσεις που έκανε. Και θα ε, ε, ήθελα να μας καλέσω όλους να είμαστε προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να κυνηγάμε διάφορες εντυπώσεις που δημιουργούνται. Ε, δεύτερον, εδώ υπάρχει ένας χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει και ένα προσαρμοσμένο νομοθετικό πλαίσιο που να απαγορεύει και να ρυθμίζει κάποιες πρακτικές που μπορεί να αποδειχθούν άκρως επικίνδυνες. Τρίτο και τελευταίο, και αυτό είναι τραγική ηρωνία, αυτός ο Κινέζος επιστήμονας ε, λέει ότι χρησιμοποίησε ως ε, τεχνική την CRISPR-Cas9 που χρησιμοποιούμε στα φυτά ενώ το απαγορεύουμε στον άνθρωπο ε,